<clears throat> Thank you very much, members. We will resume today's business with the last point, number seven on today's agenda. το τελευταίο σημείο, 7, ενίσχυση της δημοκρατίας της Μολδαβίας. Βοήθεια προς τη χώρα. Σχέδιο γνωμοδότησης από τον συγκεκριτή της Άλντε. Μικροοικονομική βοήθεια για δημοκρατία της Μολδαβίας, πρώτας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 100 εκατομμύρια ευρώ για τη Μολδαβία που τη μορφή δανείων και χορηγιών γνωρίζουμε ότι διαπιστώθηκε το 2014 απάτη οι ηγέτες της Μολδαβίας και πρώην Πρωθυπουργός τσέπωσαν ένα δισεκατομμύριο ευρώ από τις διαφορετικές τράπεζες. Μετά το σχηματισμό ενός κυβερνήσεως, σε συμφωνία με το Δούνε του, Ξαναστέλουμε ενισχύσει από το Δεκέμβριο 2016 προ τη Μολδαβία. Δίνουμε και άλλη οικονομική βοήθεια σωστή ρήξη του προπολογισμού. Την γνωμοδότηση θα συμβάλλουμε στην έκθεση τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου που θα ψηφιστεί στι 25 Απριλίου. Η συγητή ζήτησε συγγνώμη, διότι δεν παραστεί σήμερα. Θα μιλήσει εκ μέρου του συνάδελφος Δησάνες από την Άλτε που θα παρουσιάσει η γνωμονοτήσεως ε, εκ μέρους του κυρία. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κ. Σασταβίτσιος είναι στην ε, Γενέβη για την 34η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΙΟΕ και ζητά συγγνώμη που δεν παρίσταται να παρουσιάσει τη θέση του όσον αφορά τη μακροοικονομική ενίσχυση της Μολδαβίας. Το είπατε προηγουμένω ότι η Επιτροπή προτείνει να δώσουμε 100 εκατομμύρια ευρώ στη Μολδαβία από τη μορφή δανείου, 60 εκατομμύρια και η μορφή επιδοτήσεων 40 εκατομμύρια γνωρίζοντα ότι ε, η τελευταία ενίσχυση μακροοικονομική φύσεω που δόθηκε την Ευρωκένωση στην Μολδαβία ήταν 90 εκατομμύρια. Ο ε, εισηγήτη θέλει να ενισχυθεί το κείμενο προ δύο βασικέ κατευθύνσει. Ε, πρώτο σημείο, θα πρέπει προφανώ να ενισχυθεί η αρχή τη δημοκρατία, οι δημοκρατικέ αρχέ. Θα πρέπει να στηριχθεί η ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου η ανεξαρτησία και ο πλουραλισμό των μέσων ενημέρωση, η καταπολέμηση τη διαφθορά που ενισχυθεί και η καταπολέμηση επίση τη απάτη. Υπενθυμίζοντα ότι αυτό θα πρέπει να καταλήξει σε μια αποτελεσματική εφαρμογή τη έρευνα όσον αφορά να εξηχνιαστεί και η τραπεζική απάτη ε, που διεπράχθη το 2014. Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει, όπως ο ο εισηγητής, να εφαρμοστούν αρχές ερεσιμότητας θα πρέπει να υπάρχουν σημεία αναφορά σαφή, θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά εκθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο και αναστολή των πληρωμών αν δεν υπάρχει διαπιστωμένη πρόοδος επί των παναφεθέντων σημείων. Α, δεύτερη κατεύθυνση που τονίζει ο εισηγητής είναι ότι θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετέχει περισσότερο στις διεργασίες, κυρίως στην προετοιμασία του, ε, του μνημονίου θα πρέπει να δίδονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την εκταμείευση της μακροοικονομικής αυτής βοηθείας. Αυτές οι πληροφορίες, λέει ο εισηγητής, θα πρέπει να διαμοιράζονται καλύτερα ε, και να ενημερώνεται πλήρως το Ευρωκοινοβούλιο. Τρίτο σημείο, ο εισηγητής ε, υπογραμμίζει ότι η κατάσταση Μολδαβία είναι ιδιαίτερα δυσχερής και λαμβάνοντας υπόψη τι επικείμενες, βουλευτικέ τις εκλογές, ε, τον Νοέμβριο του 2018 είναι προς όφελος Ευρωπαϊκής Ενώσεως να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις παρέχοντας αυτή την ενίσχυση στις προτινόμενες προθεσμίες. Άρα θα ήταν σωστό να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες 2017 του 2018, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν όροι πιο αυστηροί ε, και προφανώς θα είναι χρήσιμος μοχλός για να υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Κλείνοντας. Ο εισηγητή σα προτείνει την υποστήριξη τη προτάσεω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσθέτοντα κάποιε εγγύσει που ανέφερα, μέτρα προστασία πιο συγκεκριμένα, πιο στεναρά, σε υπόψη ε, τις εξελίξεις στο δημοκρατικό περιβάλλον στην ε, Μολδαβία. Ε, θέλει να ευχαριστήσει του και όλους και ο εισηγητής για τη συνεισφορά του, Θα ακουστούν άλλωστε και συνημερώνει ότι η συνεδρία των σχεδόν εισηγητών θα διοργανωθεί την κατά τη εβδομάδα για να τα λήξουν αυτοί στις κατάλληλες συμβαστικές λύσεις. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Κουμπατσέλη δεν είναι εδώ. Κρίστη εκ μέρου του ΕΛ και σκιώδε εισηγητέ μα δηλαδή τώρα. Παρακαλώ. Ναι, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι Μολδαβοί και οι αρχέ και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ενθάρρυνσης και στήριξης σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αν δούμε τις μεταρρυθμίσεις και το χάρτη πορείας, η συμφωνία με το Δουνουτού και η έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων από τον Επίτροπο Χάν και την ύπατη ε, εκπρόσωπο Μογκερίνη, προφανώς έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και η στήριξή μας αυτή θα είναι ένα νέο σημείο κίνηση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα το δεύτερο εξάμεινο του 2017. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύ. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Μα γι' αυτό και δεν υπογράφουμε λευκή επιταγή, αλλά βάζουμε κριτήρια, όρου και προϋποθέσεις και στόχου που πρέπει να υλοποιηθούν. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια ευρώ που μειώθηκαν όμως σε 1 εκατομμύριο τελικά. Οι επιχορηγήσεις από 50 εκατομμύρια μειώθηκαν σε 40 εκατομμύρια και η χρηματοδότηση θα εγκριθεί μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί προϋποθέσεις πλήρως θα υπάρξουν συγκεκριμένα κριτήρια για την εκταμείευση κάθε τμήματος, γιατί η πληρωμή θα γίνεται τμήματικά και το κάθε τμήμα θα εκταμιεύεται μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, έτσι όπως αναφέρονται στο μνημόνιο το οποίο επισυνάπτεται. Τέλος, αγαπητοί συναδελφοί, ναι, αυτή η μακροοικονομική συνδρομή θα αντιμετωπίσει τι ανάγκες της Μολδαβία, αλλά δεν πρόκειται μόνο για αυτό. Πρόκειται για ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που δείχνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τη δημοκρατία της Μολδαβία. Με την συνδρομή αυτή θα έχουμε ένα παραπάνω επίπεδο πίεση προς τη χώρα για να τηρήσει του στόχου σύμφωνα με την ε, συμφωνία όπως την ανέφεραν οι συνάδελφοι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής τώρα, εκ μέρους του ΙΣΙΑΡ, κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι η μικροχρηματοδοτική ενίσχυση είναι πολύ σημαντική για τον λαό της Μολδαβίας και έχοντας μάλιστα υπόψη και την προηγούμενη εμπειρία και ιδίως την εκτεταμένη διαφθορά Είμαστε υποχρεωμένες να έχουμε υπόψη τον ειδικό μηχανισμό και ιδίως την αναστολή εν τέλει της χρηματοδότησης σε περιπτώσεις τέτοιες. Ανησυχώ ωστόσο για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μολδαβία. Αναφέρομαι σε δικηγόρους και υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων. Νομίζω επίσης ότι η Μολδαβία γίνεται όλο και περισσότερο ένα πεδίο δράσεως των ρωσικών στρατηγικών επικοινωνιών. Και λόγω ενός μονοπωλίου στην πράξη σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία μέσων μαζικής ενημέρωσης, το οποίο οφείλει να ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση στην ύπατο εκπρόσωπο να ενισχύσει έτσι περαιτέρω τις προσπάθειές της για να βελτιώσει τις επιχειρησιακές ε, δυνατότητες της Stratcom East. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγκα. Δεν βλέπω άλλους και οδησυγητές, λέει ο Προεδρεύων κύριος Μακάλιστερ. Βλέπω ωστόσο την κυρία Χάρμς που έχει ζητήσει να λάβει το λόγο. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσέλθει η σκιώδη μας και την αντικαθιστώ. Συμφωνώ με τη γνώμη που εξέφρασε η κυρία Φωτίγκα ότι σημειώνονται προβλήματα στη Μολδαβία και στο πλαίσιο των ρωσικών στρατηγικών τις οποίες χαρακτηρίζω ως αντιευρωπαϊκές. Θέλω όμως να προσθέσω ότι στη Μολδαβία βλέπουμε και εσωτερικά προβλήματα ε, που ας πούμε παράγονται επιτόπου από αυτούς που προσπαθούν να ανακτήσουν την επιρροή υπέρ της Ρωσίας στη Μολδαβία και γι' αυτό εκφράζω την ικανοποίησή μου για τις τροποποίησεις, τις τροπολογίες που έχουν γίνει και που αναφέρονται στις διάφορες ιδέες σχετικά με την αποπολιτικοποίηση των ε, διορισμών σε δημόσιες υπηρεσίες, επίσης μιας προσπάθειας επίτευξης ουδετερότητας και αυτονομίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και για την ε, λειτουργία των χρηματοδοτικών μηχανισμών μας, για την επιμονή στην διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς στην Μολδαβία, καθώς επίσης και ειδικότερα σε αυτή την τεράστια υπόθεση της τραπεζικής κλοπής. Εδώ και χρόνια ασκούμε πίεση προς την κατεύθυνση μιας δικαστικής έρευνας, αλλά δεν βλέπουμε πρόοδο. Μαζί με την πολιτική μου ομάδα είμαι υπέρ της χρηματοδοτικής στήριξης της Μολδαβίας, ταυτόχρονα όμως είμαι υπέρ του να καταστεί πιο ορατή η κριτική μας στάση καθώς και οι παρατηρήσεις μας σχετικώς με αυτά που θεωρούμε ότι δεν πάνε καλά στην Μολδαβία και ιδίω ό,τι αφορά τις ε, αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας αυτής. Ευχαριστώ αγαπητή Ρεμπέκα Χάρμς. Ο κύριος Ζόριν Μόιζερ που είναι ο εισηγητής της Επιτροπής Εξωτερικού εμπόριο, διεθνούς εμπόριο καλύτερα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ο κ. Μωυσά. Μιας και είμαι ο εισηγητής της αρμόδιας για το νομοθέτημα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Έχω ακούσει τις ανησυχίες των συναδέλφων σας που τείνουν να προτείνουν κατά κάποιο τρόπο ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική αιρεσιμότητα που έχουμε συνδέσει με τον παρόντα μηχανισμό. Οι δε ανησυχίε απηχούνται και στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους της Επιτροπής Εξωτερικών. Το πρώτο ζήτημα που θέτω είναι η φύση του μηχανισμού. Πρόκειται για μακροοικονομική ενίσχυση, IMF type, που ε, στηρίζει την, ε, το ισοζύγιο πληρωμών συνδέεται με την οικονομική διακυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί στο είδος προϋποθέσεων που μπορούμε να επιβάλλουμε στην μακροοικονομική χρηματοδότηση, διότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες στήριξης από πλευρά Ένωσης, όπου εκεί μπορούν να μπουν περισσότεροι όροι αιρεσιμότητας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εδώ θα περιοριστούμε απλώς στην αιρεσιμότητα της μακροοικονομικής Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροφή έχει θέσει υπόψη και των χωρών μελών και των τριών εισηγητών του Κοινοβουλίου ένα μη έγγραφο που περιλαμβάνει τα όσα θεωρεί ότι πρέπει να αποτελούν τη δομή τη μελλοντική συμφωνία με τη Μορδαβία. Οι πιο πολλέ ανησυχίε μα απηχούνται στο κείμενο αυτό και μάλιστα με έντονε διατυπώσει και μάλιστα με έναν τρόπο που είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στο πραγματικό κόσμο. Δηλαδή αγώνα κατά τη διαφθορά και του πλησίματο βρώμικου χρήματο, ε, αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, της διοίκησης, η FC8, εκτός από την ερεσιμότητα για την ε, μακροοικονομική στήριξη. Αυτά έχουν ένα συστημικό χαρακτήρα και εφόσον γίνουν σωστά έχουν συστημική απόδοση και μειώνουν για παράδειγμα την δύναμη των ολιγαρχών και οποιαδήποτε αυθαίρετη ε, δύναμη, διότι ε, μειώνοντας έτσι τη δύναμη των ολιγαρχών και τα λοιπά, μειώνεται και τη δυνατότητα αυτών να επηρεάσουν τη δημόσια ζωή. Και αυτό ανταποκρίνεται σε μια από τις ε, σημαντικότερες ανησυχίες που απηχούνται από τις τροπολογίε. Έλαβε επιστολή του Επιστρόπου Μοσκοβισή σήμερα, ο οποίος επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων την αυστηρή κρίση των προϋποθέσεων που θα γίνει πριν από την ε, χρηματοδότηση, πριν από τη χωρί χρηματοδοτήσεω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο θέμα, η πρόταση βασίζεται σε διαθεσμική συμφωνία, η οποία ισχύει από το 2013, ενώ μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών θεσμών. Τώρα βεβαίω είναι πιο περίπλοκο το θέμα, αλλά δεν έχω τόσο χρόνο. Αν προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε σε βάθο την συμφωνία αυτή και πολλέ από τι τροπολογίε τη Επιτροπή σα θα οδηγούσαν σε τροποποίηση τη συμφωνία πλαισίου. Αυτό όμω θα οδηγήσει σε σημαντική καθυστέρηση η οποία καθυστέρηση θα στείλει ασφαλώς το λάθος γεωπολιτικό μήνυμα και στη Μονταβία και στους ανατολικούς γειτονές μας. Είχαμε τη δυνατότητα διότι για δύο χρόνια δεν υπήρχε MFA assistance, διότι τα τρία θεσμικά όργανα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν πώς είναι καλύτερο να γίνει. Και το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεως αυτής είναι τελικό το πλαίσιο το οποίο απηχείται πιστά στην απόφαση που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξυλώσουμε αυτή την ευαίσθητη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμών. Όλοι θέλουμε ε, να βελτιωθεί η κατάσταση στη Μολδαβία. Όμως να βάλουμε όρου που σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όλα τα πράγματα μέσα σε λίγους μήνες, που ούτε καν οι χώρε μέλη δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιου υψηλέ απαιτήσει. Σημαίνει στην ουσία ότι αρνούμεθα στη χώρα αυτή την αναγκαία χρηματοδότηση. Και αν επιμείνουμε σε άλλο ε, είδου μηχανισμό, δεν θα έχει την απαραίτητη, την αναγκαία μάλλον ε, επίπτωση. Στήριξη λοιπόν της Μολδαβίας για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Εγώ μάλιστα έλαβα διαβεβαίωση από τον Επίτροπο και κλείνω κύριε Πρόεδρε, από τον Επίτροπο Μοσκοβισή, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει ακριβώς την ίδια ενημέρωση και στον ίδιο ακριβώς χρόνο όπως οι χώρες μέλη, η Επιτροπή χώρας, ε, των χωρών μελών Δηλαδή οι ανησυχίε των συναδέλφων μα σχετικά με την μη ενημέρωσή του δεν θα ισχύουν πλέον διότι έχουμε γραπτή δέσμευση από τον Μοσκοβισή ότι θα ε, ενημερώσει πλήρω το Κοινοβούλιο. Βεβαίω, όπω λέμε στα αγγλικά, το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Χρειάζεται ερεσιμότητα, υπάρχει ερεσιμότητα, χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Βεβαίω θα τη συζητήσουμε και με του άλλου ηγητές και με του κοιόδης ένα ισχυρό πακέτο αιρεσιμότητας το οποίο θα προκαλέσει πραγματικές αλλαγές αλλά με ρεαλιστικό τρόπο. Δηλαδή με μια βάση ρεαλιστική και όχι στη βάση μιας ουτοπίας και με πλήρη σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους, συγητή και σκιώδους συγητής, σκησιτές της Επιτροπής σας, καθώς και μόνο τους υπολείπους συναδέλφους, για να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Με την ελπίδα να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το κείμενο στην Ολομέλεια του Μαΐου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ κύριε Μουίζα. Ευχαριστούμε για το μας είπατε εκ μέρου τη ΣΥΝΤΑ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο συνάδελφο που θέλει να παρέμβει στη συζήτηση αυτή, οπότε θα δώσουμε το λόγο τώρα στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προηγουμένως όμως, να σας ενημερώσω ότι έχουμε καλέσει και το ελεγκτικό συνέδριο για να μας παρουσιάσουν τα δικά τους συμπεράσματα μετά την τελευταία έκθεση που είχε να κάνει με την ενίσχυση της δίκησης στην Μολδαβία. Δεν ε, μπορούσαν να έρθουν όμως, αλλά θα σας αναφέρω κάποια στοιχεία από την έκθεσή τους αυτή που έχουν σχέση με τα όσα συζητάμε. Λοιπόν, εκτίμησαν κατά πόσο 782 εκατομμύρια ευρώ που πήγανε από το 2007 στην Μολδαβία συνεισέφεραν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της δημόσιας δίκησης. Κλείνει η παράθεση από την έκθεση. Το συμπέρασμα είναι ότι η χρηματοδότηση αυτή συνεισέφερε περιορισμένα και ότι δίκες θα μπορούσε να ανταποκριθεί πιο γρήγορα. Σημειώνει επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τι προποθέσει κάθε φορά που εκταμιεύει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν αρκετά αυστηρή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αξιολόγησε επαρκώ κατά πόσο οι προποθέσει είχαν καλυφθεί όχι. Τώρα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών και ίσως θα μπορούσαν να σχολιάσουν και τι έκαναν σε σχέση με την έκθεση αυτή του ελεγκτικού συνεδρίου και πώς ανταποκρίθηκαν στις παρατηρήσεις αυτές προκειμένου η βοήθειά μας στη Μολδαβία να είναι πιο αποτελεσματική στο μέλλον. Ποιος? Ο κύριος Ελαιοδόρου Τεμπράνο Αρόγιο, σωστά? Ωραία. Παρακαλώ, είσαστε επικεφαλής του Τμήματος για την Μακροοικονομική Συνδρομή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Στροβίτσο, τον εισηγητή, και τον κύριο Μόισα, τον εισηγητή εκ μέρους της ΣΥΝΤΑ, για την πρόταση αυτή. Όπως γνωρίζετε, η Μολδαβία έχει περάσει από μία περίοδο μακροοικονομικής ε, συνδρομής από το 2002 εξαιτία διαφόρων προβλημάτων που είχε τραπεζική κρίση, για παράδειγμα μετά από μια μεγάλη απάτη και δέχασε και τη στήριξη σε ένα βαθμό από διάφορους εταίρους Ρωσία κτλ. Έχει λοιπόν αυτή την συνδρομή μεταξύ άλλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση διεκόπη μέχρι να αναλάβει νέα κυβέρνηση στην αρχή του 2016 και υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες σιγά σιγά εφαρμόζονται. Μεταρρυθμίσεις που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που οδήγησαν τον Φεβρουάριο που μας πέρασε και σε ένα χάρτη πορείας με κατά προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις. Στη συνέχεια υπήρξε ε, συμφωνία και με το Δουνουτού για ένα ε, πρόγραμμα μαζί τους, το οποίο άρχισε να υλοποιείται. Το δούνο του λοιπόν είναι στη χώρα. Ε, ολοκληρώνεται ικανοποιητικά η πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος αυτού. Και αρχές Απριλίου θα το εγκρίνει ε, το δούνο του. Συνεπώς υπάρχει εδώ πέρα ένα άνοιγμα θετικό που μπορεί να βοηθήσει η βοήθειά μας, η οποία όπως σας είπα διακόπη για δύο χρόνια. Έχουμε την μακροοικονομική αυτή συνδρομή και στα πλαίσια αυτά προτείνουμε τη συνδρομή αυτή, αλλά πρέπει να είμαι απόλυτα σαφής ότι συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ευρωβουλευτές εδώ. Όσον αφορά την αιρεσιμότητα, τις προϋποθέσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να είναι αυστηρή με την προσέγγιση αυτή βάση προϋποθέσεων, εκταμείευση βάση κριτηρίων και προϋποθέσεων, ήδη από την αρχή, από τα πρώτα τμήματα της εκταμείευσης και θα υπάρξει και backloading που θα είναι ένα βασικό στοιχείο της συμφωνίας αυτής. Κυκλοφόρησε ένα non-paper, όπως ο κύριος Μόση, που επικεντρώνεται σε διάφορες μεταρρυθμίσεις κλειδί. Ένα εγκάρσιο ζήτημα είναι η ενίσχυση της διακυβέρνησης, της οικονομικής, της δημοσιονομικής, της τράπεζας, στο δημόσιο τομέα, με εξωτερικούς οικονομικούς ελέγχους, ε, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες προμήθειες. Και ένας άλλος τομέας θα είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομοποίησης παράνομου χρήματος. Ένα άλλο στοιχείο ενίσχυσης της διακυβέρνησης είναι και η διασυνδεσιμότητα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τελευταίο, το κλίμα επενδύσεων με το SFTA. Αυτό ε, συνδέεται γιατί οτιδήποτε διακόψει την διαδικασία που θα ήταν για παράδειγμα διακοπή του FCDA θα ήταν πρόβλημα, αλλά και επειδή έχουμε συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις όσον αφορά την συμφωνία της EFT. Όπως είπε και ο κύριος Μόισεν, δεν περιμένουμε η μακροοικονομική συνδρομή να λύσει όλα τα προβλήματα ε, σε σχέση με τη χώρα αυτή και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται. Η συνδρομή αυτή θα εξαρτάται από την υλοποίηση τέτοιων μεταρρυθμίσεων. Βάζουμε δηλαδή τέτοιες προϋποθέσεις που είναι οικονομικής, δημοσιονομικής υφής, αλλά έχει να κάνει και με θέματα διακυβέρνησης και με μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα που θα επηρεάσουν το επενδυτικό κλίμα. Σας διαβεβαιώ, όπως συμβαίνει πάντα, πριν γίνει οποιαδήποτε εκταμείευση ή πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, θα χρειάζεται αξιολόγηση και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αν υπάρχουν προβλήματα πολιτικά ή σχετικά με τους δημοκρατικούς θεσμούς ή με την διαδικασία σύνδεσης κτλ. Όλα αυτά θα οδηγούν σε διακοπή της συνδρομής. Εμεί προτείνουμε καταρχήν το 40% της συνδρομή. Πρόκειται για μια πολύ φτωχιά χώρα, αν λάβουμε υπόψη μας στου διάφορους δείκτες. Χρέος και Και είναι και η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει τη συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που σημαίνει ότι συνθέτει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας επιτρέπουν να αποφασίσουμε για τη συνδρομή αυτή. Υπογραμμίζω επίσης ότι πολλές από τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου καθησυχάζονται από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε στην δράση συνδρομής. Το μνημόνιο και η δημοσιονομική συμφωνία περιλαμβάνει εγγυήσεις προστασίας οικονομικών συμφερόντων για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα, ότι θα επιτρέπονται έλεγχοι από την ε, όλα, το ελεγκτικό συνέδριο κλπ. Έχουμε και κάποιες διατάξεις οι οποίες όχι απλώς διακόπτουν την εκταμείευση έτσι και υπάρχει παραμικρή παρατυπία, αλλά θα υπάρξει πλήρης διακοπή. Συνεπώς, όπως συμβαίνει και με το Δουνουτού, αν υπάρξει διακοπή των μεταρρυθμίσεων ή όχι επαρκής πρόοδος, δεν θα υπάρξει ούτε εκταμίευση. Οι συνομοθέτες εγκρίνοντας την ε, συμφωνία αυτή για τη συνδρομή δεν σημαίνει ότι επιτρέπει και τις εκταμιεύσεις. Όχι, απλώς επιτρέπει την χρήση του εργαλείου αυτού της μακροοικονομικής συνδρομής και εφόσον υπάρξει καλή πρόοδος, τότε θα υπάρξει και εκταμίευση. Και βάσει των ε, προτάσεων τροποποίησης που περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση, τις τροπολογίες δηλαδή που υποβλήθηκαν, νομίζω ότι είναι σημαντικό να περιορίσουμε τις τροπολογίες. Γιατί, όπως υπόθηκε ήδη, οι μακροοικονομικοί κανόνες απορρέουν από δύσκολους και λεπτούς συμβιβασμούς τους οποίους κατέληξαν οι συνομοθέτες πριν από τρία χρόνια στην ε, κοινή δήλωση για την μακροοικονομική συνδρομή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λοιπόν, υπάρχει κίνδυνος για την ισορροπία αυτή αν τεθούν υπό οι κανόνες οι οποίοι αποφασίστηκαν τότε. Βέβαια, οι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως και του Συμβουλίου αντικατοπτρίζονται πολύ καλά εφόσον κάνουμε πιο σκληρή τη γλώσσα όσον αφορά τις προϋποθέσεις που συνδέουμε με την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων κτλ. Η αιρεσιμότητα μέσα σε αιτιολογικέ σκέψεις μπορούμε να αναφέρουμε πιο πολύ το μνημόνιο, τις προϋποθέσεις, ότι η Επιτροπή έχει την εντολή για διαπραγματεύσεις κτλ. Άρα, σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Αναφέρομαι και στην ε, πρόσφατη ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Επιτρόπου μας στον πρόεδρο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώνει πλήρως το Κοινοβούλιο βάσει της κοινή δήλωσης των συνομοθετών, αν πρόκειται για εκταμιεύσεις, αν πρόκειται για μνημόνια, αν πρόκειται για επιτροπές που μπορεί να δημιουργηθούν, επιτροπολογία. Το μνημόνιο αμέσως θα πάει στο Συμβούλιο και την και το Κοινοβούλιο. Και αν υπάρξει εκταμίευση, για κάθε δόση της εκταμίευσης και η αξιολόγηση που θα συνοδεύει την εκταμίευση αυτή είναι πράγματα τα οποία θα φτάνουν αμέσως στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ό,τι άλλη πληροφορία μπορεί να θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γραπτά ή αν θέλετε να έρχεται η επιτροπή στις συνεδριάσεις σας, ευχαρίστως θα ανταποκριθούμε για να σας ενημερώνουμε πλήρως με ό,τι πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό λέει και η επιστολή του Επιτρόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Ρόγιο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σούμπελ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε να απευθυνθώ στο κρατήριο εδώ. Να αναφερθώ στην πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία. Είδαμε κάποια σταθερότητα να επικρατεί τον τελευταίο χρόνο περίπου. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση και νέο πρόεδρο από το τέλος Δεκεμβρίου παρελθόντος έτους. Ο κ. Δοντών, ο πρόεδρος, επέστρεψε από δεύτερη επίσκεψη στη Μόσχα, όπου προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι εύκολο. Τούτου λεχθέντος. Παρά τη σταθερότητα, η Δημοκρατία της Μολδαβίας αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα, πολλά από αυτά ήδη αναφέρθηκαν από τους προλαλήσαντες. Κυρίως πρέπει να καταπολεθεί η διαφθορά και έχουμε και προβλήματα διακυβέρνηση. Άρα και η οικονομική θέση και οι πληρωμές έχουν αποδυναμωθεί και επίσης η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Επόμενα προβλήματα, όπως αναφέρθηκε, είναι να διαλευκανθεί η απάτη, η τεράστια που έπληξε την οικονομία της χώρας το 2014. Μας είπαν τη δεύτερη έκθεση της Αμερικανικής εταιρείας Kroll που δημιουργεί τον έλεγχο δημοσιευτεί τον Απρίλιο. Ελπίζουμε αυτή η έκθεση να διαφωτίσει το ζήτημα και όπως είπε η κυρία Χάρμ τελικά να δώσει αποτελέσματα. Και πορίσματα σε αυτή την έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του πολιτικές πολιτικέ εξελίξει στη Μολδαβία. Αναφέραμε ότι θα θέλαμε να δούμε συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Φεβρουαρίου 2016. Όλα αυτά τα συμπεράσματα, όσα συμπεριλαμβάνονται, ισχύουν μέχρι σήμερα. Κάποια οικονομικά προβλήματα αυξήθηκαν λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και των σχέσεων τη Μολδαβία με εμπορικούς εταίρου τη. Αυτό εξορροπήθηκε από αύξηση εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνια συνδεση Σύνδεσης από 1η Ιουλίου 2016 ετέθησε ισχύ. Εδώ και μια εβδομάδα, 13 Μαρτίου, δημοσιεύθηκε μια έκθεση για την εφαρμογή τη Συμφωνίας Σύνδεση με τη Μολδαβία και αναφέρεται η πρόοδο για την εφαρμογή τη συμφωνία σύνδεση και τη δημιουργία ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Και αναφέρονται ποιε μεταρρυθμίσει πρέπει να γίνουν. Θα τα συζητήσουμε στην, στο επικείμενο Συμβούλιο Σύνθεσης, 31 η Μαρτίου. Ο Πρωθυπουργό Φίλιπ τη μονταβιας θα παραστεί. Θα προεδρεύει η υπατο εκπροσωπο η κυρία Μογκερίνη. Προτείνεται μακροοικονομική βοήθεια τη ευρωπαικη ενωσεω και θα συνοδεύει το πρόγραμμα του Δούνου του για τη χώρα. Συμφωνήθηκε αυτό πέρσι τον Νοεμβρίο. Οι εκταμιεύσει σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση τη μορφών τη χώρα με το πρόγραμμα του Δουνουτού και ότι θα εφαρμόζουν διάφοροι όροι της πολιτικής. Αντικείμενο συμφωνίας του μνημονίου μεταξύ Μολδαβίας, της Δημοκρατίας Μολδαβίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτοί οι όροι θα προσπαθούσαν να καλύψουν τις αδυναμίες της οικονομίας της χώρας και αδυναμίες του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης και του τραπεζικού τομέα. Θα υπάρξει στενό συντονισμό με τα προγράμματα που έχει συμφωνήσει με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα η Δημοκρατία της Μολδαβίας. Και σύμφωνα με τους άλλους όρους που έχει ε, συμφωνήσει η χώρα. Οι όροι για τη στήριξη της οικονομίας στην πλευρά Ευρωπαϊκή Ονίσου δεν εξαρτώνται από τα θέματα της ανεξαρτησίας του δικαστικού τομέα και της καταπολεμήσεως της διαφθοράς. Η Μολδαβία μπόρεσε να εφετήσει κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις στους τελευταίους μήνες Τώρα όμως πρέπει να συνεχιστούν τα βήματα αυτά και πρέπει να ενισχυθούν χωρίς υπαναχωρήσεις. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε να εξυγχρονιστεί η χώρα. Αυξήθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές και οι επαφές μεταξύ των λαών. Πιστεύουμε ότι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Να βοηθήσουν τη, βόρα, τη χώρα να δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες. Διότι υπάρχουν δυνατότητες εμπορίου και τεχνογνωσία που μπορούμε να δώσουμε στη χώρα. Μπορούμε να δώσουμε και προοπτικές στους νέους της χώρας για να εργαστούν. Συνοψίζοντας, θέλουμε να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τη χώρα στις μεταρρυθμίσεις που προσπαθεί. Αλλά όπως αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2016, περιμένουμε απτά αποτελέσματα. Υπό αυτούς τους όρους υποστηρίζουμε ε, αυτή την πρόταση για μακροοικονομική ενίσχυση της Μολδαβίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σούμπελ, συνάδελφοι. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια μήπως. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Ένας, δύο, δύο συνάδελφοι. Η κυρία Χάμς πρώτη. Νομίζω ότι όλοι μας, εμείς που θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα, για όλους μας είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο λαός της Μολδαβίας περιμένει να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τα τεκτενόμενα. Τι γίνονται τα χρήματα που δίνουμε. Περιμένει ο λαός της Μολδαβίας να μην είμαστε συνένοχοι εκείνων που χρησιμοποιούν τις δομές που επικρίνουν πολλοί πολίτες της χώρας. Όχι μόνο εδώ τις επικρίνουν. Όχι μόνο το ελεκτικό συνέδριο και εμείς επικρίνουμε τις δομές, αλλά και πολλοί πολίτες της Μολδαβίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη Συμφωνία Σύνδεση πρέπει να το λάβει αυτό. Είναι κρισίμου σημασία να το λάβει αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεσαγνέ. Να ευχαριστήσω εν ονόματι του εισηγητού. Θα διαβιβάσουμε προφανώ τα υποθέτα. Κυρίω αυτά που μας συνάδελφοι τη ΑΦΕΤ και τη ΣΥΝΤΑ Υπάρχει συνένεση ουσιαστικά. Για τη μακροοικονομική βοήθεια, ότι στέλνουμε θετικό ισχυρό μήνυμα προς τη Μολδαβία. Υπάρχει και άλλη συμφωνία ότι πρέπει να επιβληθούν όροι οικονομικοί ορθής διακυβέρνησης που προχωρούν παράλληλα. Το είπαν και συνάδελφοι Τσίντα. Πρέπει να είναι ρεαλιστικοί όροι και απαιτητικοί προς όφελος και των δύο πλευρών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Μολδαβίας. Αυτά είχα να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουμε ξανά μια παρέμβαση του κ. Μόιζερ. Α, ένα σχόλιο σε αυτά που είπε η κυρία Χάρμς. Συμφωνώ. Περιμένει ο λαός τη Μολδαβία να γνωρίζουμε πού πήγαν τα χρήματα. Σε αυτή την περίπτωση και αυτό το μέσο είναι εύκολα τα πράγματα. Τα χρήματα θα πάνε στην Εθνική Τράπεζα. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένου σκοπού. Ένα σκοπό. Την υποστήριξη του ισοζυγίου πληρωμών. Τα χρήματα δεν πάνε σε προγράμματα κάποιου ολιγάρχου και να μπορεί να τα επεξαιρέσει. Μιλάμε για μακροοικονομική βοήθεια που βεβαίω δεν σημαίνει ότι για άλλα μέσα θα πρέπει να εξετάζουμε πραγματικά που πηγαίνουν τα χρήματα. Εδώ ο κίνδυνος να δαπανηθούν λάθος τα χρήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτος και έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα προληπτικά ούτω ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά μιλούμε για μακροοικονομική ενίσχυση, δεν μιλάμε για χρηματοδότηση προγραμμάτων. Κανεί δεν μπορεί να τα υπεξαιρέσει. Κλείνοντα, πρόκειται για ένα κομμάτι ευρύτερη εικόνα χρησιμοποιούμε μόχλευση μεταρρύθμισης για τη Μολδαβία. Και προστατεύεται αυτή η προσέγγιση από καταχρήσεις και παρεμβάσεις. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα μέσα ενισχύσεως που δίνουμε στην Μολδαβία ότι έχουν πραγματικά αντιχτυπώ υποφθυρούς όρους. Και αυτή η αιρεσιμότητα είναι στο πακέτο δεν είναι εφημισμός ο ρεαλισμός για δυναμία. Όχι, το πακέτο ερασιμότητας που ετοιμάζεται είναι κάτι ισχυρότατο. Και αν λειτουργήσει θα έχει συστημικά αποτελέσματα πάρα πολύ σημαντικά. Σε σημαντικότατη κλιμάκα. Αυτά έχω να πω και ευχαριστώ. Καλώς. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, Ευρωπα... της Επιτροπής, ε, συγγνώμη, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής και τους συναδέλφους για τη συζήτηση. Τελικά, να πω πότε θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την 11η Απριλίου, Πέμπτη. Και έχουμε χρόνο πριν διαβηχώρα ψηφοφορία στην Επιτροπή Ιντε, που θα γίνει στις 25 Απριλίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά για σήμερα νομίζω. Η επόμενη συνάντησή μας, αύριο το πρωί, 8 και 30 το πρωί. Θα γίνουν μία-δύο ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα σημεία 8, 9, 10 και θα συνεχίσουμε στις 8.45 ανταλλαγή απόψεων με τον Άνταμ Σαμπ, θα το γνωρίζουν περισσότερο από εσά. Επιτετραμένος της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, της, των Ηνωμένων Πολιτείων στις Βρυξέλλες. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.